Okay, colleagues. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη, το σχέδιο. Μπορούμε να την εγκρίνουμε. Πολύ ωραία. Τώρα η χρόνη συζήτησης είναι λίγο χαλαρή δεν θα τους στηρίσουμε πιστά. Ε, έχουμε και την αυριανή ψηφοφορία. Κάποια στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάποια διακοπή. Γιατί έχουμε πάνω από 200 τροπολογίες. Παρά τις συμβαστικές τροπολογίες και τους ε, συνδυασμούς που θα γίνουν. Θα ξεκινήσουμε πάντως όπως προβλέπετε σε νέα. Αλλά χρειαστεί να κάνουμε κάποια διαλύματα. Επόμενο θέμα, λεπτομέρειε τη επίτευξη του στόχου μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Το 2020. Η συντάκτρια της γνωμοδότηση είναι η κυρία Γκαρδιασάβαλ Ρουμπιάλ. Έχετε το λόγο κυρία Συγγετρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω εν συντομία την κατάσταση. Όπως είπατε, έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα είχαμε γύρω στις 80 τροπολογίες, για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα λίγο λιγότερες. Στην πρώτη συζήτηση επί των δύο γνωμοδοτήσεων έγινε σαφές ότι υπήρχε αρκετή διάσταση απόψεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων και μάλιστα αυτή η διάσταση έλαβανε ε, μεγάλες διαστάσεις σε ορισμένα σημεία και με σχετικά γεφύρωτες διαφορές. Πάντως ε, συνεργάστηκα με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα ε, συνεδριάσαμε οι σκιώδεις ηγητές προσπαθώντας να συγκλίνουμε τις απόψεις. Μάλιστα εξετάσαμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες που υπέβαλα προς τις πολιτικές ομάδες την προηγούμενη εβδομάδα και μάλλον υπάρχει κάποια απάρχη συμφωνίας. Αν και στο μεταξύ προέκυψαν και άλλες διαφορές και μια και είναι πολύ σημαντική συζήτηση με μεγάλη απόκληση στην αρχή βαίνουμε προς μια σύγκληση, αλλά δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει τις συμβαστικές τροπολογίες. Πάντως ευελπιστώ ότι σήμερα το απόγευμα οι σκιώδεις ηγητές ε, θα συνεχίσουν τη συνεργασία μαζί μου προκειμένου να διευκρινίσουμε τα εκρεμή ζητήματα που δεν είναι καν ε, λεπτομεριακά, είναι σημαντικά, ώστε αύριο όταν κληθούμε να ψηφίσουμε για τις δύο να έχουμε καταλήξει στη συμφωνία. Και τα λέω αυτά γιατί θα είναι κρίμα να μην καταλήξουμε συμφωνία. Έτσι θα χάσουμε την ευκαιρία να τροποποιήσουμε, έστω και μέσω μιας γνωμοδότησης, την ε, έκθεση της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος που έχει κοινή δερμοδιότητα με την Επιτροπή Βιομηχανίας για το θέμα αυτό. Αλλά θεωρώ ότι και εμείς θα πρέπει να υποβάλουμε τη γνωμοδότησή μας και να ασκήσουμε κάποια επιρροή. Έχουν απομείνει όμως εκκρεμεί κάποια σημαντικά θέματα, όπως είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος, αν θα έχουμε ποσοτικοποιημένο στόχο, έστω και ενδεικτικό, για μετά το 2020, για το 2025 δηλαδή. Και επίσης το θέμα των υπερμορίων, άλλο σημαντικό ζήτημα. Το θέμα των υπερμορίων είναι σημαντικό. Εγώ έχω υποβάλει εναλλακτική πρόταση ως προς τα πιστοτικά υπερμόρια που θεωρώ ότι ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα και μπορεί να βοηθήσει και τη βιομηχανία να υλοποιήσει τους νέους στόχους και θεωρώ ότι είναι και πιο δίκαιη η πρόταση για τα πιστοτικά υπερμόρια. Δυστυχώς όμως δεν είναι της ίδιας γνώμης οι πολιτικές ομάδες. Γι' αυτό και άλλαξα τη συμβαστική μου τροπολογία ως προς το θέμα αυτό, επιδιώκοντας μία συνεννόηση με τους οι υπόλοιπους συναδέλφους. Πάντως να κρεμεί κάποια αρκετά σημαντικά ζητήματα και θα ήθελα να σας θέρμο παρακαλέσω να καταβάλουμε όλοι κάποια προσπάθεια. Γιατί ναι, δεν υπάρχει διάσταση απόψεων, αλλά νομίζω ότι έχουμε την υποχρέωση, την ηθική υποχρέωση να καταλήξουμε σε συμφωνία για να βελτιώσουμε με τη γνωμοδότησή μα την έκθεση τη επιτροπή, των αρμοδίων επιτροπών. Στην Επιτροπή Βιομηχανία, επίση διαπιστώθηκε μεγάλη διάσταση απόψεων, αλλά παρόλα αυτά τελικά όλες οι πολιτικές ομάδες με αμοιβέ υποχωρήσεις και εμένοντα σε κάποια στοιχεία κατέληξαν σε συμβαστικές τροπολογίες. Ελπίζω και στη δική μας Επιτροπή να καταφέρουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία, ώστε αύριο να υπερψηφίσουμε την γνωμοδότησή μας, της Επιτροπής Μεταφορών δηλαδή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φλόρεντ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η συνεργασία μας. Ακόμα και αν είχαμε επιμέρους διαφωνίες, ε, στόχος όλων ήταν στο τέλος να καταλήξουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα και για το περιβάλλον αλλά και για τα αυτοκίνητα και με ρωτήσετε και εμένα, ακόμα και για τα γρήγορα αυτοκίνητα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και οικονόμοι και φιδωλοί. Λοιπόν, σύντομα να επικεντρωθώ στο συμβιβασμού. Το, πρώτο μας βρίσκει σύμφωνο ε, και με χαρά υπερψηφίζουμε. Ο δεύτερος συμβιβασμός μας προβληματίζει. Έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ακόμα να τον υπερψηφίσουμε. Δεν ξέρω μήπως αλλάξει η διατύπωση ε, για να το ξανασυζητήσουμε γιατί έχετε και δύο αριθμούς. Αν ε, αναφερθεί ρητά ότι δεν είναι δεσμευτική αυτή. Αυτό το προτείνω ε, για να έχουμε πιο μεγάλη συνοχή τελικά και συνέχεια στο κείμενό μας. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να βγούμε έτσι θαραλέα και να πούμε ότι θέλουμε 65 το 2025. Ξέρω ότι ορισμένοι συνάδελφοι το επιθυμούν, αλλά κάποια στιγμή αυτά που λέμε θα πρέπει να είναι εφικτά και υπολογίσιμα. Να ανοίξουμε μια κατεύθυνση, να δείξουμε το διάδρομο, όχι με καταληκτική ημερομηνία και καταληκτικό ε, αριθμό. Να το ξανασυζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη συμβαστική τροπολογία παριθμών 3, με χαρά να την υποστηρίξουμε αν εκτός από τα 2,5 γραμμάρια προσθέστηκε ε, μία ένδειξη ετησίως. Συμβιβαστική τροπολογία παριθμών 4 με τον κύκλο δοκιμής το δεχόμαστε και το συμβιβαστικό 5 με τον κύκλο ζωής επίσης. Το ίδιο ισχύει και για τα ημιφορτηγά, τα λεγόμενα επαγγελματικά και σταματώ εδώ. Σήμερα το πρωί ήρθα το αυτοκίνητο σε ε, μια μεγάλη διαδρομή από την εκλογική μου περιφέρεια μέχρι τις Βρυξέλλες και είδα ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι τα ορυκτά καύσιμα ε, στα αυτοκίνητα ε, είναι πεπερασμένα προφανώς. Γι' αυτό θέλουμε αυτοκίνητα τα οποία να ε, είναι οικονομικά και να υπάρχουν αυτοκίνητα και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Λοιπόν, μόνο αν είμαστε θαραλέοι ε, στη νομοθεσία μας, τότε θα έχουμε ακόμα καλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία, πράγμα που είναι όνειρό μου. Ευχαριστώ για την Άλντε Μπιλμπάου. Ευχαριστώ. Απουσιάζει ο αρμόδιος για το θέμα αυτό, αλλά μου ζήτησε να σας μεταφέρω τη θέση του για την γνωμοδότηση. Καταρχήν, ως προς τις διαφορές για τις εγκρίσεις τύπου και την κατάσταση στα, στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, διαφέρουν ε, οι εκπομπές αυτές από τις πραγματικές. Και μάλιστα έχουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα ανάλογα με τη θερμοκρασία. Η μηχανία επιλέγει την καλύτερη, την πιο βολική λύση, ώστε να καταλήξει σε χαμηλές τιμές διοξιδίου του άνθρακα. Δεύτερο θέμα, σε ό,τι αφορά τους στόχους για το 2020. Η ε, κυρία Μέισνερ, ε, η σκιοδησηγητρία, θεωρεί ότι η συγγήτριά μας προτείνει στόχους για μετά το 2020 μεταξύ 65 και 75 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα για τα επιβατηγά και 100 με 115 γραμμάρια το χιλιόμετρο για ελαφρά ε, φορτηγά. μετά, ε, βέβαια, η κυρία Μέισνερ θεωρεί ότι δεν θα συμφωνήσει με τους στόχους για μετά το 2020 δεδομένου ότι προτείνει ποσοτικοποιημένους στόχους για το 2025. Ούτε το, την ψαλίδα δέχεται η κυρία Μέισνερ, γιατί ουσιαστικά δεσμεύει την αυτοκινητοβιομηχανία και θεωρούμε ότι και τους στόχους για το 2015 θα πρέπει να τους δούμε αργότερα σε μια νομοθετική πρόταση. Σε ό,τι αφορά για τους στόχους μετά το 2015, η κυρία Μέισνερ θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, ως σημείο αναφοράς η συμβαστική λύση της Επιτροπής Βιομηχανίας ε, που συγκέντρωσε μεγάλη πλειοψηφία στην ψηφοφορία. Και τώρα σε ό,τι αφορά τα πιστοτικά υπερμόρια, όπως ε, και για το θέμα των στόχων για μετά το 2020, η κυρία Μέισνερ προτείνει καταλληλότερη λύση την συμβαστική τροπολογία της Επιτροπής Βιομηχανίας με ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από το 2016 θεωρώντας ότι ε, το όριο το 2,5 γραμμαρίων ισχύει για κάθε χρόνο. Ο κύριος Τέιλορ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που προσπάθησε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν είχαμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερη, ιδιαίτερα πετυχημένη συνάντηση συντονιστών. Υπήρξε μια ανταλλαγή ισχυρών επιχειρημάτων, προσπαθήσαμε να βρούμε κοινοτόπο θα έλεγα, αλλά κάποιες από τις λεγόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες στις οποίες συμπεριελήφθηκε και το όνομά μου σε ορισμένες από αυτές, ενώ η δική μου τροπολογία ήταν ακριβώς η αντίθετη από αυτό το οποίο ζητούσε η συμβιβαστική. Θα ζητήσω λοιπόν από το όνομά μου να αποσυρθεί από κάποιες από τις τροπολογίες αυτές. Μιλώντας γενικότερα τώρα, την ίδια, το ίδιο δεκαπενθήμερο όπου η Volkswagen ξεκίνησε ένα υβριδικό αυτοκίνητο ενός λίτρου το οποίο εκπέμπει 24 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα. Όταν βλέπουμε λοιπόν το δρόμο που μας δείχνει η βιομηχανία και μας λέει η βιομηχανία ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα καλύτερο από το 147 για τα φορτηγάκια και 97 για τα αυτοκίνητα, ε, τώρα δεν θα πρέπει και να τους πολυπιστεύουμε. Νομίζω ότι στόχος των διακανονιστικών ρυθμιστικών αρχών είναι να προσπαθήσουμε να καθοδηγήσουμε την πρόοδο και δυστυχώς δεν το έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Το θέμα μας είναι λοιπόν εμείς να πρωτοπορούμε και όχι να αντικατοπτρίζουμε τις πιο συντηρητικές αντιλήψεις που πρεσβεύει η βιομηχανία των αυτοκινήτων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πράγματι οι αυτοκινητοβιομηχανίες κερδίζουν τεράστια ποσά και οι εκκλήσεις τους και τα παράπονά τους για τη μεγάλη τους φτώχεια είναι κούφια λόγια. Θα υποστηρίξουμε την εισηγήτρια λοιπόν όπου αυτό είναι εφικτό και θα αποσύρω βασικά το όνομά μου από κάποιες από τις συμβιβαστικές, λεγόμενες συμβιβαστικές. Ευχαριστώ κύριε Τόιλορ. Ελπίζω να πιείτε και καφέ. Όπου, όπου να είναι θα έρθει. Μπορεί ο κύριος με τον καφέ να πάω στον Τέιλορ αντί να πάει ο Τέιλορ στον καφέ. Ροσμπάχ. Θα είμαι πάρα πολύ συνοπτική. Η ομάδα μας συμφωνεί με τις θέσεις της συζητήτριας. η στόχη είναι φιλόδοξη και εφικτή για την βιομηχανία. Τουλάχιστον έτσι μας λένε. Οι στόχοι για τις εκπομπές θα πρέπει να εξυπηρετούν τον σωστό τρόπο για την μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 με σημαντικό τρόπο. Έχουμε λοιπόν ε, μια συζήτηση να κάνουμε για το τι θα συμβεί για μετά το 2020 ή 2025. Εμείς συμφωνούμε με τους νέους κύκλους ελέγχου σαν πιο θετικούς για τον καταναλωτή. Θα πρέπει να μειωθεί το κενό ανάμεσα στις θεωρητικές εκτιμήσεις και στην πραγματική κατανάλωση. Τώρα για τα λεγόμενα πιστοτικά υπερμόρια. Ε, νομίζω λοιπόν ότι σε σχέση με αυτά τα πιστοτικά credits ε, έχουμε ακόμα ε, πολύ δρόμο να κάνουμε. Ο κύριος Κόλιτσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι εκπομπές καυσαερίου και η μείωση μάλλον των εκπομπών καυσαερίου είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος και θα πρέπει να τον επιδιώξουμε μεν τον στόχο αυτό, αλλά η επιδίωξη αυτή θα πρέπει να γίνει μέσω της βελτίωσης των συνθήκων, των μεθόδων και των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε διάφορες παραμέτρους όπως την κατάσταση των ελαστικών, τη ρύθμιση του κινητήρα αλλά και το ύφος οδήγησης γιατί μόνο και μόνο με την αλλαγή του στυλ οδήγησης ε, αν οδηγούμε φυσιολογικά και γαλήνια και όχι σαν οδηγία αγώνων θα κερδίσουμε πάρα πολλά σε σχέση με τις εκπομπές καυσαερίων. Είναι αλήθεια ότι ορισμένα οχήματα, σε ορισμένες χώρες μάλιστα, και αναφέρομαι στη Γαλλία και σε κάποιες άλλες χώρες, είναι σε τόσο κακή κατάσταση που φοβάται κανείς ότι θα ξεκολλήσουν κομμάτια από αυτά τα σαράβαλα που κυκλοφορούν σε χώρες σαν τη Γαλλία. Πέραν τούτου συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι οι κανόνες που πρέπει να δημιουργήσουμε θα πρέπει να είναι σεβαστοί. Δεν ξέρω αν ο στόχος θα είναι 95 ή 70 για το αλλά νομίζω ότι οι τεχνικές προϋποθέσεις εξαρτώνται εν πολλής από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το όχημα. Τακτική λοιπόν έλεγχη τεχνική των αυτοκινήτων και αστυνομική έλεγχη τακτική των αυτοκινήτων θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι θα πετύχουμε σημαντικές βιώσεις, ε, μειώσεις της εκπομπής χωρίς πάρα πολλές επενδύσεις. Θα πρέπει βέβαια να δούμε τι θα κάνουμε και σε τομείς οι οποίοι απαιτούν επενδύσεις όπως η προώθηση της τεχνολογίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ένας τρίτος δρόμος είναι τα, ε, αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με υδρογόνο. Είναι κάτι όμως το οποίο εδώ απαιτεί χρόνο αλλά είναι κάτι το οποίο τεχνολογικά θα συμβεί, όχι στο έβδομο πλαίσιο βέβαια. Η έκθεση λοιπόν που έχουμε μπροστά μας είναι σημαντική, αναφερόμαστε στις εκπομπές διοξιδίου ε, στη συγκεκριμένη φάση για τα ελαφρά φορτηγά, αλλά δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών. Εκεί έχουμε πάρα πολλά κενά στην νομοθεσία μας και οφείλουμε να επανέλθουμε. Υποστηρίζω λοιπόν λέει ξανά ο κύριος Κόχλητς εκ την έκθεση αυτή αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί υιοθετώντα συμβιβαστικές προτάσεις όπως αυτές τις οποίες αναφέρθηκε ο συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και το δικό μας όδη εισηγητή. Το θέμα βεβαίως δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι επί της ουσίας, παρόλο που στη σύνολη πολιτική μεταφορών αντιμετωπίζουμε ε, πολύ αυτά τα ζητήματα. Ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η μείωση του διοξυνδίου του άνθρακα για μας είναι και παραμένει ε, σημαντική και αναπόφευτη. Έχουμε μάθει και από το παρελθόν ότι αν είναι απλώς εθελούσια αυτή η ρύθμιση δεν πετυχαίνουμε το στόχο μας. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βεβαίως και για μας αλλά και για πολλούς συναδελφούς εξακολουθεί να ισχύει ότι βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίες από παντού. Από τη μια η τεχνολογία περιγράφεται περίπου ανέφικτη, αυτή που ζητούμε, ενώ κάποιοι άλλοι λέγουν ότι είναι κάλλιστα εφικτή. Εάν βρούμε ένα σωστό νομοθετικό δρόμο θα πρέπει να αναζητήσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Εμείς ως ΕΛΚ συμφωνούμε, όπως προηγουμένως εξήγησε ο Καλχάιντς Φλόρενς, με τη γραμμή αυτή. Σε ό,τι αφορά ε, το κύκλο δοκιμών και τους καταναλωτές, θα πρέπει ο καταναλωτής να είναι σωστά ενημερωμένος για να μπορεί να κάνει και σωστά τις δοκιμές. Με σωστή πληροφόρηση και καλή ενημέρωση. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν ανταποκρίνεται ε, στην πραγματικότητα. Είναι μεροληπτική και περιορισμένη ενημέρωση. Θα πρέπει να τα γνωρίζει όλα ε, ο ο καταναλωτής. Σε ό,τι αφορά τα υπερμόρια της super credits, προέρχομαι από μια χώρα εγώ που ε, ε, έχει ε, προχωρήσει σε περικοπές ορισμένων κινήτρων για λόγους οικονομίας. αυτά είναι ημίμετρα. Εγώ προτιμώ να παραμένουν τα κίνητρα παρά να έρχονται κυρώσεις εκ των υστέρων. Σε ό,τι φορά τους στόχους μετά το 2020, δίστανται απόψεις. Πολύ ωραία τα εξήγησε ο Φλόρενς. Ε, ορισμένοι λέγουν ότι ε, χρειάζονται ε, από τώρα τιμές συγκεκριμένε, άλλοι λέγουν όχι μετά το 2016. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς το ΕΛΚ είναι ότι πρέπει να ξέρει η βιομηχανία ότι μετά το 2020 θα πρέπει να κάνει περαιτέρω προσπάθειες. Αν αυτές θα είναι από τώρα ποσοτικές και καθορισμένες είναι άλλη ιστορία. Ε, πάντως την κατεύθυνση θα πρέπει να τη δώσουμε. Επίσης ζούμε σε χώρες Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία ε, έχει και κάποια οικονομική αξία για την οικονομία των χωρών μας. Ε, αυτά όλα λοιπόν που είναι πάρα πολύ δεσμευτικά και πιεστικά θα πρέπει να ε, μπορούν να συγκεραστούν με την οικονομία, με τη βιομηχανία και τις θέσεις εργασίας. Και από την Ένωση να δείξουμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι μεταφορές στους δεσμευτικούς στόχους ε, για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε και από αλλού. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένους τομείς, αλλά όχι μόνο στις μεταφορές να γίνονται περικοπές. Αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε. Νομίζω θα ήταν καλύτερο να λάβουμε υπόψη μας και άλλους κλάδους της οικονομίας. Ε, είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε διάφορες συμβαστικές προτάσεις, τα είπε ο κύριος Φλόρενς και ελπίζω να ε, καταλήξουμε σε μια ε, ισχυρή φωνή από την Επιτροπή Μεταφορών. Ο κύριος Ελχαντράουι. Ευχαριστώ Πρόεδρε ακούω πολύ ε, ε, με χαρά να ακούω τους συναδέλφους ότι είναι υπέρ ε, της πρώτης αυτής. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστική η προσέγγιση της ΣΕΙΔΕΡ, της συγκήτριάς μας. Προσπαθεί με πολύ λογικό τρόπο να αντιμετωπίσει ένα θέμα περίπλοκο σαν αυτό που αντιμετωπίζουμε. Ελπίζω ειλικρινά η Επιτροπή Μεταφορών να μπορέσει να στείλει ένα χειρό μήνυμα με μεγάλη πλειοψηφία να υποστηρίξει τις προστάσεις της. Στην Επιτροπή Ήτρε, ας πούμε, κατέστη δυνατό κάτι τέτοιο, είναι ενωμένη. Ε, σε ό,τι αφορά τις δοκιμές συμφωνώ, θα πρέπει να ε, προσαρμοστούν οι μέθοδοι και να ε, συνάδουν με τα όσα μπορεί κανείς να αναμένει σε φυσιολογικές συνθήκες. Καταλαβαίνω ότι γίνεται τώρα μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθούν νέε μέθοδοι και νέε διαδικασίε. Αλλά εμεί τι θα πρέπει να κάνουμε, περιμένουμε να ολοκληρωθούν αυτέ οι διαδικασίε και να δώσουμε μόνο μία ένδειξη, μία κατεύθυνση στην αυτοκινητοβιομηχανία για τους στόχους τους πιο μακροπρόθεσμους. Έχω την αίσθηση ότι εδώ διήστανται οι απόψεις μας. Η συγγήτρια έχει κάνει μια πρόταση πάρα πολύ καλή δεν έχει συγκεκριμένους στόχους. Μια ψαλίδα προτείνει ένα φάσμα για να μπορεί να εργάζεται και η αυτοκινητοβιομηχανία. Δείχνει απλώς την κατεύθυνση ε, μακροπρόθεσμα γιατί ε, για να αναπτυχθεί ένας νέος τύπος, τύπος αυτοκινήτου χρειάζεται χρόνια. Θα πρέπει να μπορεί να προσανατολιστεί η αυτοκινητοβιομηχανία για το νέο κύκλο δοκιμών και να κανονίσει την πορεία της. Αλλιώ μπορεί να είναι πολύ μικρό το διάστημα που τη δίνεται για να προσαρμοστεί. Αυτό τα λέγω για να σας καλέσω να κοιτάξετε την τροπολογία της εισηγήτριας και να ε, καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Σύντομα λοιπόν ως πολιτική ομάδα εμείς υποστηρίζουμε την εισηγήτριά μας και ελπίζουμε για αύριο να υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία, όχι μόνο γι' αυτό και για άλλα θέματα. Κάπου πρέπει να βρούμε τη μέση λύση. Καταλαβαίνω ότι οι πράσινοι δεν είναι πλήρω ικανοποιημένοι, ούτε η Άλντε ούτε το ΕΛΚ, αλλά δεν μπορούμε η Επιτροπή μας να, στείλουμε ένα μήνυμα επιτέλους ε, ότι ε, κάτι προτείνουμε και συμφωνούμε με αυτό όλοι. Ο κύριος Ρικέ, ευχαριστώ. Καταρχήν, θερμά ευχαριστώ προς την εισηγήτρια και να πω ε, παραθέσει ότι ως μέρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, έχω πρόβλημα με τους αριθμούς. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς τους γενικούς στόχους, αλλά όταν αρχίζουμε και μετράμε κατά λεπτό σε γραμμάρια ή μήνες ή χρόνια, τα πράγματα περιπλέκονται. Συμφωνώ πάντως με τη γνώμη του συντονιστή μας, του κυρίου Γκρός, ότι θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των διστάμενων απόψεων και των ενισχυλιών του καθενός. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Η 31η Δεκεμβρίου 2014 Ω καταληκτική προθεσμία για τις μελέτες και την υποβολή των νέων στόχων είναι ουτοπική. Είναι αδύνατο μέχρι το τέλος του επόμενου έτους να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα στοιχεία που χρειάζεται και ταυτόχρονα να κάνει τις μελέτες και να προσδιορίσει τους στόχους για μετά το 2020. Νομίζω θα πρέπει να αφήσουμε λίγο χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην την πιέσουμε, γιατί δεν θα προλάβει. Δεύτερη παρατήρηση. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ μεταξύ ε, όσων ε, ε, είναι υπέρ της μείωσης των εκπομπών, δηλαδή όσοι έχουν μεγάλες οικολογικές ευαισθησίες, ε, ενώ ταυτόχρονα δεν θέλουν να ενθαρρύνουν, να παρατηρούν την αυτοκινητοβιομηχανία να κάνει προσπάθειες. Οπότε καλό θα ήταν τα πιστωτικά υπερμόρια να αυξηθούν αντί να μειωθούν, να θέλουμε ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα που να λειτουργούν με υδρογόνο ή μπαταρίες. Αν περιοριστούμε στο όριο το 1,3 γραμμάρια δεν θα δώσουμε ουσιαστικά κίνητρα στην μηχανία για να προχωρήσει. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα να ε, μαστιγώνουμε το άλογο για να προχωρήσει και να τραβάμε τα χαλινάρια ή θα δώσουμε κίνητρα να προχωρήσει με ε, ναύσματα ε, στην αυτοκινητοβιομηχανία και με αντίστοιχα πιστοτικά υπερμόρια για να μπορεί να προσαρμοστεί. Γιατί και τα 20.000 αυτοκίνητα είναι ελάχιστο αριθμό. Αν θέλουμε κάποια στιγμή περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ υψηλότερων πιστοτικών υπερμόριων. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να καλωσορίσω και μία αντιπροσωπεία από το Ίδρυμα Φρέντερικ Ιμπεκ από τη Γερμανία. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ελπίζω να θεωρήσετε χρήσιμη και ενδιαφέρουσα την επίσκεψή σας. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Κολουμπιεύσκα. Να απαντήσω στα τρία βασικά θέματα που συζητήθηκαν σήμερα. Στόχοι 2020, κύκλος ελέγχου και ε, πιστώσεις, τα λεγόμενα super credits. Εμείς προωθούμε τη συλλογή δεδομένων διαφορετικού τύπου πολύ περισσότερο από ότι τώρα για μετά το 2014. Κάποιες μελέτες έχουν ξεκινήσει προπαρασκευαστικά. Είναι δυνατόν να πετύχουμε τους στόχους του 20 λοιπόν. Οι στόχοι του 95 ε, γραμμαρίων για την προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί έχει οδηγήσει σε μια σημαντική μείωση των εκπομπών επιβατηγών αυτοκινήτων για τον κύκλο ελέγχων δοκιμασιών. Η νέα διαδικασία τεστ, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από το 2014 και σε πλήρη εφαρμογή το 2017, θα ελέγχει πολύ καλύτερα, πληρέστερα τις ε, <clears throat> εκπομπές καυσαερίων. Αυτό είναι κάτι στο οποίο έχει επιμείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και γενικότερα όλοι οι εμπλεκόμενοι. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Και τέλος, σε σχέση με τα super credits. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία εδώ, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή κινητήρων <clears throat> με χαμηλές ε, ε, εκπομπές καυσέριων είδαμε ότι οι προτάσεις που γίνονται στις τροπολογίες δεν <clears throat> δημιουργούν κάποιες χρονικές προθεσμίες για την απόσυρση των παλιών τεχνολογιών κτλ. Και δεν θέτουν και το θέμα της συζήτησης για το τι θα γίνει μετά το 2020 ή 2025. Εμείς εξηγήσαμε στο μη έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της θέσης μας και ελπίζουμε να το χρησιμοποιήσετε σαν βάση για τις συζητήσεις που θα κάνετε από εδώ και πέρα. Η συγήτρια. Ευχαριστώ. Όπως διαπιστώσατε και από τη συζήτηση, υπάρχει διάσταση, πολύ μεγάλη διάσταση απόψεων. Για να μην πω ότι έχουμε τόσους απόψεις όσο και μέλη στην Επιτροπή Μεταφορών. Και τα πιο επίμαχα σημεία, όπως ακούσαμε, είναι τα πιστοτικά υπερμόρια, οι στόχοι μετά το 2020, αλλά και το θέμα της έγκρισης τύπου ε, για τις εκπομπές, για τους κύκλους δοκιμών και να προσαρμοστούν αυτές οι εκπομπές με τη πραγματικότητα. Είχαμε πάντως συμφωνία σε κάποια επιμέρους σημεία και μερικές από τις τροπολογίες αυτές και μια συμβαστική τροπολογία ακολουθούν αυτή την πορεία. Σε ό,τι αφορά τους στόχους για μετά το 2025. Νομίζω ότι υπάρχουν επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ και των δύο απόψεων. Και οι δύο θέσεις είναι λογικές και με μια τροπολογία μου εγώ προσπάθησα να βρω μια χρυσή τομή. Γιατί ναι, μεν υπάρχει μεγάλη ακόμη αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθούν οι νέες τεχνολογίες ό,τι αφορά τη μείωση πομπών διοξιδίου του άνθρακα και γίνονται νέες δοκιμές. Αλλά ταυτόχρονα είναι αλήθεια ότι αν δεν, ήδη, δεν αρχίσουμε ήδη να επεξεργαζόμαστε νέους στόχους για το 2025, ίσως α, ε, μας ξεπεράσουν τα γεγονότα και οι εξελίξεις. Γιατί η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία μα είπε ότι χρειάζεται τουλάχιστον μία επταετία για να προβλέψει για τα αυτοκίνητα τα επιβατικά και τουλάχιστον δέκα για τα επαγγελματικά. Οπότε αν καθυστερήσουμε με τους νέους στόχους του 2025 η αυτοκινητοβιομηχανία πολύ εύλογα και δικαιολογημένα θα πει ότι δεν προλαβαίνει να εφαρμόσει τις νέες διαδικασίες που χρειάζονται για να υλοποιήσει τους νέους στόχους. Γι' αυτό λοιπόν ε, Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένο αριθμό. Γι' αυτό και πρότεινα εγώ ένα φάσμα, μια ψαλίδα εκπομπών. Και με όλα τα στοιχεία που έχουμε, θεωρούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο στόχο για το 2015 θα κοιμαθεί μεταξύ των 65 και των 75 γραμμαρίων για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Οπότε έκρινε σημαντικό και θεωρώ ε, σημαντικό να δώσουμε μια κατεύθυνση ε, και το μήνυμα μας υπέρ της ε, μείωσης των εκπομπών του άνθρακα και να δώσουμε και μια πορεία προς την αυτοκινητοβιομηχανία για να ξέρει τι κατεύθυνση να ακολουθήσει. Θα συνεχίσουμε βέβαια ε, την εξέταση των προτάσεων με τις πολιτικές ομάδες, αλλά στόχος μας είναι να δώσουμε ε, ένα μήνυμα και μια κατεύθυνση για το προς τα που θέλουμε να κινηθούμε. Άλλωστε ο στόχος είναι ανοιχτός και τα... οι τιμές αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Νομίζω από μόνο το αυτό είναι σημαντικό. Το θέμα είναι ότι αν όλοι εμείνουμε πεισματικά και αμετακίνητοι στις θέσεις μας, παρόλο που είναι εύλογες, τότε δεν πρόκειται να καταλήξουμε πουθενά. Θα πρέπει όλοι να κάνουμε προσπάθειες και υποχωρήσεις για να βρούμε μια συμφωνία. Γιατί καλύτερα να έχουμε μια συμφωνία από ότι να μην καταλήξουμε πουθενά και να ε, μείνουμε στην θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμετάβλητη. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστοτικά υπερμόρια. Θέλουμε να βοηθήσουμε τη βιομηχανία και να δώσουμε αυτή την επιβράβευση ή αυτή τη βοήθεια για τη συνέχιση της ε, καινοτομία και της έρευνας και της πώληση ηλεκτρικών ε, οχημάτων ή υβριδικών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ως προς τα πιστοτικά υπερμόρια μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Για παράδειγμα να πούμε ότι είναι το ανώτατο όριο 2,5 γραμμάρια ετησίω. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε εκεί. Και τώρα πότε θα αρχίσουν να λειτουργούν ή πότε λήγουν τα πιστοτικά υπερμόρια θα το συζητήσουμε αργότερα ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέχρι αύριο το πρωί. Κύριε Τέιλορ, σε ό,τι αφορά τι συμβαστικέ τροπολογίε, το κατά πόσο οι δικέ σα τροπολογίε καλύπτονται από τι συμβαστικέ τροπολογίε. Νομίζω ότι είναι λάθος αντίληψη οι δικέ μου τροπολογίε, οι τροπολογίε μάλλον που εγώ ανέταξα στι συμβαστικέ τροπολογίε, καλύπτονται σε αδρές γραμμέ, Δεν καλύπτονται όλες διεξοδικά. Σε μερικές τροπολογίε καλύπτω κάποιε προτάσει των πρασίνων και αναφέρω δεικτικά ποιες τροπολογίε πάνω κάτω καλύπτω. Κύριε Ρικέ, σε ό,τι αφορά την 31η ε, Δεκεμβρίου του 2014. Σε μια συμβαστική τροπολογία έχουμε αναβάλει και το 2015 αυτή την προθεσμία, γιατί θεωρούμε ότι ο Δεκέμβριος του 2014, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θεωρεί ως εφικτό στόχο, εμείς κρίνουμε ότι παρά είναι φιλόδοξος και πολύ κοντινός. Γι' αυτό και προτείναμε παράταση μέχρι το 2015. Υπάρχουν προτάσεις για το 2017 ή 2018, αλλά τότε είναι υπερβολικά αργά για την αυτοκινητοβιομηχανία, γιατί η αυτο, αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι στην τελική ανάλυση αυτή που θα κληθεί να υλοποιήσει τους στόχους. Επαναλαμβάνω πάντως ότι είμαι διαλλακτική και πρόθυμη να συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις με τις ομάδες και θα δούμε αν αύριο καταλήξουμε σε συμφωνία οριστική που θα αποκρισταλώνει και θα διευκρινίζει τη θέση της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για τα επιβρατιά αυτοκίνητα θα γίνει 24 ή 25 και για τα ελαφρά φορτηγά την 6η και 7η Μαΐου. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η στρατηγική για την αηφόρο κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μάικλ Κρέμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ, κύριο Κράμερ. Είναι μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλούμαστε εμείς ως Κοινοβούλιο να διδράσουμε. Η ανακοίνωση έχει το τίτλο «Έρευνα και καινοτομία για τη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη, χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη τεχνολογία των μεταφορών». Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδης ηγητές. Ήταν καλή η συνεργασία όσο και η ανταλλαγή απόψεων και ορισμένα από τα επιχειρήματα ε, τα έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου. Είναι πολύ ευρεία ε, η βάση συνεργασίας λοιπόν. Ε, την έχω χωρίσει την έκθεση σε τρία μεγάλα κεφάλαια. Ε, γενικές αρχές πρώτα, γενικά μέτρα στη συνέχεια και ακολουθούν τα ειδικά μέτρα. Βεβαίως θέλω να πω εδώ ότι και η έκθεση της Κομισιόν είναι καλή από μόνη της, αλλά ξέρουμε ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Και ως Κοινοβούλιο είμαστε πάντα πεπισμένοι ότι ποτέ δεν επιδεινώνουμε την έκθεση, πάντα τη βελτιώνουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δούμε τι θα βγει όμως και από το τελικό αποτέλεσμα. Γενικές αρχές το πρώτο. Τι λέμε εκεί δεν κοιτάμε ένα χρονικό διάστημα, αλλά ένα ε, κύκλο ζωής, ας πούμε, στα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Όταν ε, ε, κινείται ένα ηλεκτροκίνητο όχημα, δεν εκπέμπει καυσαέρια προφανώς, αλλά θα πρέπει να δούμε σε όλο τον κύκλο της ζωής του γενικότερα τι εκπομπές έχει. Και επίσης η τεχνολογική ουδετερότητα συμφωνήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Να ε, ε, το καθορίσουμε από την αρχή γιατί πρόκειται για έρευνα και καινοτομία. Αν τα ξέραμε όλα δεν θα τα χρειαζόμασταν αυτά τα κείμενα. Τεχνολογική ουδετερότητα λοιπόν μας ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα και επίσης δεν θέλουμε μόνο να κοιτάμε τι κάνουν οι μεγάλες εταιρείες και οι μεγάλοι όμιλοι, θα πρέπει να λειτουργούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και από πλευράς εθνικής οικονομίας έχει αυτό σημασία, αλλά όχι μόνο. Γιατί η καινοτομία ξέρετε ότι προέρχεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θυμάμαι ακόμα τους πρώτους ηλιακούς ε, συλλέκτες και τις πρώτες ανεμογεννήτριες ήταν ε, ορισμένοι εφευρέτες που τα κάναν στα γκαράζ τους και όλοι τους περιγελούσαν. Και τώρα είναι η τεχνολογία του μέλλοντος. Ποτέ δεν θα είχε ασχοληθεί ένας μεγάλος όμιλος. Μικρομεσαίοι είναι αυτοί που καινοτομούν, που ψάχνουν, που ερευνούν και έχουν και την ελευθερία να το κάνουν σε αντίθεση με τους μεγάλους ομίλους. Δεύτερο κεφάλαιο, γενικά μέτρα. Βεβαίω ξέρουμε ότι ε, κάθε καινοτομία, κάθε ε, νεοτερισμός ε, είναι σημαντικός τεχνολογικά, αλλά δεν φτάνει, δεν αρκεί η τεχνολογία για το μέλλον, χρειάζεται και αλλαγή νοοτροπίας. Και εδώ Καλείται ο κάθε άνθρωπος ε, να αντιδράσει, πώς οδηγεί, ε, πώς κυκλοφορεί, τι συγκοινωνίες χρησιμοποιεί. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτόμαστε όχι πώς πάμε από το α σημείο στο β ή από ένα σταθμό στον άλλο σταθμό, αλλά πώς πας πόρτα-πόρτα. Οι Ελβετοί το κάνουν πολύ ωραία. Ε, ε έχουν χαράξει ένα αυτοκινητόδρομο, σκέφτονται ε, πώς θα, βελτι... πώς θα... ένα σιδηρόδρομο μάλλον, πώς θα βελτιωθούν 70 γραμμές στη Γερμανία, ούτε καν τα διανοούνται αυτά, απλώς σκέφτονται τα συμφέροντα της Deutsche Bahn και του κράτους. Ε, ε, ο κατώτατος μισθός παίζει όρια, παίζει, παίζει ρόλο, υπάρχουν 20 κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν βασικό μισθό, στη χώρα μου ακόμα δεν υπάρχει, ελπίζω μετά τις επόμενες ευρωεκλογές να γίνουν 21 αυτές οι 20 χώρες. Βεβαίω. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την αιωλική ενέργεια, την ηλιακή... Ε, ακόμα και όταν εφευρέθηκε ε, ε, το, η ε, ορισμένοι ε, γελούσαν για το πώς θα μειωθεί, πώς θα αυξηθεί η ταχύτητα της ναυσιπλοείας, αλλά τελικά έκανα την ανάγκη τους φιλοτιμία και προχώρησαν σε καινοτόμες λύσεις. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε και το ποδήλατο και τους πεζούς. δεν λέω το ποδήλατο επειδή είμαι εγώ ποδηλάτης, αλλά ένας πάρα πολύ συντηρητικός υπουργό μεταφορών στη Γερμανία, βαβαρός κιόλα, ε, που ε, δεν έχει γυαλιά, έχει παρμπρίζ για να κοιτάει. Αλλά αυτός λέει ε, το 90% της πόλης των αποστάσεων που κάνουμε με αυτοκίνητο είναι λιγότερο από 6 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να κάνει κανείς με το ποδήλατο, με τα πόδια η Κοπενχάγη ε, είναι θαυμάσιο παράδειγμα. Στο Αμστερντάμ είναι 31% η κυκλοφορία με ποδήλατα. Στη Δε αυξήθηκε κατά 300% μέσα σε 20 χρόνια. Αυτό είναι το μέλλον. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε το μοναδικό κοινοβούλιο στον κόσμο που έχει ε, στις εγκαταστάσεις του ε, σταθμό. Έχουμε και ένα γραφείο ειδικό για την κινητικότητα. Και αν είχαμε και τρένο για το αεροδρόμιο, το οποίο υποτίθεται ότι είναι έτοιμο εδώ και χρόνια, απλώς δεν έχουν δρομολόγια, ε, τότε ε, δεν θα χρειαζόμαστε και αυτοκίνητα για να πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο και τρεις φορές ε, λιγότερο θα διαρκούσε η διαδρομή αυτή. 12% εξοικονόμηση ενέργεια έχουμε ε, και 42% ε, στα τροχέα ε, εάν υπάρχει όριο μέσα στις πόλεις 30 χιλιόμετρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει προτείνει εδώ και χρόνια, το είπαμε και στον κύριο Κάλλας, τι αποτέλεσμα είχαμε, μηδέν στο πηλίκο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους κοιότητες ηγητές Ε, ε, συστήματα ATM, ε συστήματα τιμολόγηση των εισιτηρίων και άλλα είναι συγκεκριμένα μέτρα που πρότειναν και ο τους. Ευχαριστώ και περιμένω τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάχ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ του κυρίου Πίρκερ ε, θα ήθελα να παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μας. Ε, κολλείεται και ζητεί συγγνώμη για την απουσία του. Ε, η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές μιλά για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πιο καθαρή κυκλοφορία και πιο ασφαλή. Αυτό χρειάζονται για να γίνουν όλα αυτά, για να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα χωρίς να περιορίζεται καθόλου η κυκλοφορία και η προσωπική κινητικότητα του καθενός ή της οικονομίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν και στις μεταφορές νέες τεχνολογίες και αυτό θα πρέπει να αποκτήσει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών ε, θα πρέπει να διέπεται από τη Λευκή Βιβλοστόχος ένα σύστημα μεταφορών με συνδυασμένες μεταφορές, επιβατικές και εμπορευματικές. Για μας ε, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Η λύση της κυκλοφορίας της πόλης, 80% των Ευρωπαίων στο μέλλον θα ζουν σε πόλεις. Και εδώ η Ευρώπη έχει τεράστιες πρόκλησεις να αντιμετωπίσει. Νέες τεχνολογίες θα πρέπει να συνεισφέρουν και να είναι σε θέση να το κάνουν. Δεύτερον, περιορισμός του θορύβου. Αυτό θα γίνει με νέες τεχνολογίες, με νέες έννοιες από την αρχή, νέο σχεδιασμό δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό. Έτσι θα δέχονται περισσότερο και οι πολίτε νέες λύσεις. Η έρευνα δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Ένα τρίτο σημείο, ε, ε, εναλλακτικά συστήματα προώθησης ε, και τεχνολογίες επικοινωνιών και συγκοινωνιών με αυτοκίνητα, οχήματα καθαρά, διασυνδεδεμένα για να μπορέσουμε να φτάνουμε καλύτερα και πιο φτηνά στο στόχο μα και πιο γρήγορα στον προορισμό μας. Νέα συστήματα επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων ε, και των στόλων ε, των μεταφορών. Τεχνολογίες ε, του μέλλοντος θα πρέπει να εξαφανίσουν τα προβλήματα που έχουμε στις πόλεις με μποτιλιαρίσματα και με τους χώρους στάθμευσης. Υποστήριξη εφιών συστημάτων λοιπόν μετακίνησης, αποτελεσματική οικονομικές αλυσίδες εφοδιαστικής. Ε, αυτό έχει μεγάλη σημασία και η οικονομική ελάφρυνση και για ιδιώτες και για τις εταιρείες. Ε, θα πρέπει να ε, υπάρχουν νέα συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης των φορτίων καθοδών. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό λοιπόν στην υπόθεση των μεταφορών ε, και θα πρέπει να προωθηθούν νέες τεχνολογίες με τεχνολογική ουδετερότητα, αυτό είναι βασική αρχή, χωρίς όμως να δημιουργεί εμπόδια για την εσωτερική αγορά. Και ένα τελευταίο, τα αποτελέσματα της έρευνας στις μεταφορές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα, να κυκλοφορούν στην αγορά και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι νέες λύσεις. Μερικά πολύ θετικά σημεία είναι το 4 για την τεχνολογική ουδετερότητα, όπως είπαμε, το 6 για μεγαλύτερη υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το 16 για ε, μεγαλύτερη ε, ανάπτυξη συστημάτων πληροφόρησης, πληρωμής και κρατήσεων. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ, κύριο Σαλκαντραουή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή μας ε, για την πρότασή του. Ζητώ συγγνώμη ξενόματος του κυρίου Λιμπεράτσκι που είναι σχεδόν εισηγητής μας. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με την πρόταση του εισηγητού, του κυρίου Κράμερ. Ε, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διασυνοριακή σύνδεση και εκεί υπάρχουν κάποιοι λείποντες κρίκοι, και τα διάφορα συστήματα ε, των συνδυασμένων μεταφορών. Να πω όμως δύο λόγια εγώ για την κοινωνική διάσταση. Στο σημείο 9 λέει ο συνάδελφος Λιβεράτση ότι υποστηρίζει και αυτή την πρόταση για τη μείωση του θορύβου, αλλά να αναπτύξουμε λίγο περισσότερο και τις ιδέες μας και σε ό,τι αφορά το σιδηρόδρομο θα πρέπει να έχουμε στόχο να έχουμε πιο ε, φτηνές, ε, φτηνές λύσεις ε, με τις νέες τεχνολογίες και με τα συστήματα πλοήγησης με δορυφόρο η έρευνα, η ανάπτυξη και η νέα τεχνολογία θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να βελτιώσει την άνεση στις μεταφορές για το κοινό. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται για να μπορούν πολύ μικρές επιχειρήσεις να έχουν ε, τη δυνατότητα να αναπτύσσουν εφαρμογές, να συμμετέχουν στην αγορά και να ε, βοηθούν στην υπόθεση των μεταφορών ας πούμε, με διάφορες εφαρμογές να βοηθούν ε, τους καταναλωτές και τους χρήστες ε, στη μετακίνησή τους από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο, σε ένα εστιατόριο, σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα ταξίδι. Όλα αυτά μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέροντα για να καταλάβουν οι πολίτες πώς μπορούν να μετακινούνται και να επιλέγουν ε, τρόπους και μέσα μεταφοράς πιο αηφόρα και πιο φιλικά στο περιβάλλον. Επίσης, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική κινητικότητα μέσα στις πόλεις. Συμφωνώ πολύ με τον εισηγητή ότι ε, μπορούμε να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά μέσα στις πόλεις. Ε, έχουμε άσκοπες μετακινήσεις, ψάχνουμε πού να παρκάρουμε ε, και μας τρώει πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχουν τρόποι να λυθεί αυτό με έξυπνο τρόπο. Ας πούμε θα μπορούμε να μοιραζόμαστε ένα αυτοκίνητο ε, με διάφορα ε, συστήματα πληροφορικής και ενημέρωση. Τέλος, η βάση αυτή είναι πολύ καλή για περαιτέρω συνεργασία και καλύτερη αξιοποίηση. Θα κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας. Πάντως γενικά ε, όλοι πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση και έχουμε τον ίδιο στόχο. Ευχαριστώ κυρία Πιλμπό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθειά του, γιατί ήδη από την πρώτη συνάντηση διαπιστώσαμε ότι συμπεριέλαβε τις, τις παρατηρήσεις μας. Συμφωνώ με πολλά επιμέρους σημεία της έκθεσης. Από τις γενικές αρχές όμως λείπει η αναφορά ότι με το έργο αυτό, με την προσπάθεια αυτή, θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών που θα είναι βιώσιμο και ανταγωνιστικό ταυτόχρονα. Και είναι πολύ σημαντικό στις γενικές αρχές να προσδιορίσουμε και τους στόχους μας. Τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη της καινοτομίας, ε, της έρευνας και του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να πρωτοστατήσουμε και να έχουμε καθαρές μεταφορές, οικολογικές, βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη δηλαδή και ταυτόχρονα να δημιουργούν αυτές οι μεταφορές νέες θέσεις απασχόλησης που θα δίνουν έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και κυρίως στις επιχειρήσεις κοινωνικής καινοτομία, για να προβάλλουν αυτές ιδιαίτερα εν μέσω της κρίσης νέα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης. Κάτι άλλο που λείπει από την έκθεση είναι η μνήμα της α, ε, μεταπληκτικής βιομηχανίας, γιατί σε αυτή την προσπάθεια καινοτομία, έρευνα, συντονισμού, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια ανταγωνιστικότητα και μια βιωσιμότητα των μεταφορών, αλλά να μην ξεχνούμε και τη μεταπιτική βιομηχανία, που είναι πολύ σημαντική και τώρα, αλλά και στο μέλλον. Επίσης, πιστεύω ότι και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια χρηματοδότηση, να τις απαλλάξουμε από την υπερβολική γραφειοκρατία και συμφωνούμε με τρεις προτάσεις. Την ανάγκη ανάπτυξης της διασύνδεσης, τη διαλειτουργικότητα και τους διασμένους τρόπους μεταφοράς πολυτροπικότητα. Είναι σημαντικά αυτά τα τρία θέματα που μαζί με την καινοτομία και την έρευνα θα μας επιτρέψουν να έχουμε πιο αποτελεσματικές μεταφορές στην Ευρώπη, πιο ολοκληρωμένες μεταφορές και πιο αποτελεσματικές, ώστε να πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα που επενδύουμε και στα κράτη-μέλη και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Από αυτές τις ε, ιδέες διέπονται και οι τροπολογίες μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηχορύπανση, σίγουρα θέλουμε μεταφορές που θα παράγει λιγότερο θόρυβο, θα ενοχλεί λιγότερο και από τις συζητήσεις που κάναμε ε, έχουμε και τις ε, προτάσεις ε, του, της οργάνωσης για τους τυφλούς που μας είπαν ότι δεν θα πρέπει να ε, εξαλείψουμε τελείως το θόρυβο από τις μεταφορές, γιατί οι τυφλοί χρησιμοποιούν αυτούς τους θορύβους για να αντιληφθούν καλύτερα ε, τα μέσα μεταφοράς. Και σε ό,τι αφορά την κατάργηση των επιπέδων θορύβου, σίγουρα η συζήτηση αυτή θα είναι πολύ χρονοβόρα. Ελπίζω να μπορέσουμε αυτές τις γενικές αρχές ε, να διαμορφώσουμε μια έκθεση που θα έχει ως πρωταρχικό στόχο, όπως είπα και στην αρχή, να εξασφαλίσει παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Κυρία Ροσπάκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αντικαταστήσω το σκιώδη εισηγητή της ομάδας μου. Η έρευνα και η καινοτομία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις νέες τεχνολογίες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του τομέα των μεταφορών, αλλά και τις αντιλήψεις οι οποίες ισχύουν στον κόσμο και έτσι θα βελτιώσουμε τη συνειδητοποίηση του προβλήματος. Αν δεν ακολουθούσουν οι πολίτες και αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, τα μέτρα που θα πάρουμε δεν θα έχουν επιτυχία. Θα στηρίξουμε λοιπόν την ουδετερότητα της τεχνολογίας. Οι πολιτικές μας θα πρέπει να είναι απόλυτα ουδέτερες σε σχέση με τις τεχνολογίες. Η έρευνα και η ανάπτυξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω ευκολότερης πρόσβασης στα κοινοτικά ταμεία και μέσω της μείωσης των διοικητικών εμποδίων ολοκληρωμένα συστήματα πληροφόρησης, ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων και πληρωμών θα πρέπει να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Αυτό έχει ζητηθεί επανειλημμένα, αλλά θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε. Μερικές φορές υπάρχουν δυσκολίες για την κράτηση των απαιτούμενων θέσεων κτλ. Πρέπει λοιπόν αυτό να ισχύσει και για τις μεταφορές με λεωφορεία. Ευχαριστούμε λοιπόν τον εισηγητή για την εργασία του. Ευχαριστούμε και τους σκιώδεις εισηγητές και ε, στοχεύουμε να συνεργαστούμε μαζί τους και στο μέλλον. Κόχλιτσεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχουν κάποια επιμέρους σημεία τα οποία θα ήθελα να δω να προστίθενται στη συγκεκριμένη έκθεση. Ίσως ο εισηγητής εδώ να παρέλειψε ορισμένα σημεία. Θα ήθελα να τον καλέσω στην πόλη μου και να ποδηλατήσουμε σε εισαγωγικά μαζί για να δει πραγματικά πώς έχει η κατάσταση. Στο σημείο 9 σαν παράδειγμα, στο τμήμα 9 μάλλον, κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων. Αυτό είναι κάτι στο οποίο εμένω και το έχω ήδη αναφέρει ιδιαίτερα για τα ελαφρά φορτηγά. Νομίζω ότι οι ρυθμίσεις εδώ είναι μηδενικής ισχύως σχετικά με τους περιορισμούς ταχύτητας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει φυσικά θετικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Απ' την άλλη πάλι αν οδηγώ πολύ αργά είμαι εμπόδιο για τη ροή της κυκλοφορίας. Τίθεται λοιπόν εδώ ένα θέμα, η εκπαίδευση, η κατάρτιση. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς πιλότος αγώνων για να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο. Αν κάποιος οδηγεί γρήγορα είναι κίνδυνος για ατύχημα και με τα εμπορικά ελαφρά φορτηγά. Λοιπόν, το ίδιο επίσης ισχύει με τους νέους οδηγούς 18 ετών. Θα πρέπει να ελέγχονται συστηματικά δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, έτσι μόνο θα μειώσουμε τα σοβαρά ατυχήματα. Τώρα για τις δημόσιες, τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Κρίσιμο θέμα. Κομβικό. Σημαντικό για τις μεγάλες ιδιαίτερα πόλεις. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικέ λεωφοριογραμμές. Υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να ορίζονται τέτοιες λωρίδες σαν παράδειγμα ελεύθερες σε περιπτώσεις ανάγκης όπως έγινε στην Πράγα κατά τη διάρκεια των πλημμυρών. <clears throat> Όσον τώρα ε, όσον αφορά στην ανακύκλωση τη λεγόμενη των τρόπων μεταφοράς, των μέσων μεταφοράς εννοεί ο μιλητής, θα πρέπει να δούμε το τι κοστίζει και οικονομικά και οικολογικά η ε, ανακύκλωση των αυτοκινήτων, όπως επίσης και άλλων μέσων μεταφοράς όπως τα πλοία. Τα πλοία ε, εξάγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και δεν αναπτύσσουμε εμείς μεθόδους για να τα ε, αποσύρουμε. Στο 19 υπάρχει περαιτέρω προσπάθεια μείωσης της εκπομπής καυσαερίων στις αερομεταφορές Νομίζω ότι αυτού του είδους οι εκπομπές δεν συμβαίνουν μόνο από τις αερομεταφορές, αερομεταφορές συγγνώμη, αλλά από τις διαδικασίες εσωτερικής ε, καύσης. Και αναφέρομαι εδώ στα θιούχα, όχι στα ανθρακούχα. Συνεπώς, σχετικά με τα λεγόμενα νοξ, λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε επιπλέον προσπάθεια και στις αερομεταφορές και γενικότερα σε όλα τα είδη μεταφοράς. Αζωτούχα. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να δώσουμε ε, κάποιες ε, επιπλέον δυνατότητες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε κάποιες καινοτόμες ιδέες οι οποίες ακούγονται δεν έχουμε μακροπρόθεσμες προοπτικές στην παρούσα φάση και πρέπει να τις βρούμε αυτές τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Thank you, Mr. Thank you to your committee and uh, your rapporteur, Mr. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε τον εισηγητή, τον κύριο Κράμερ και τους σκιώδης εισηγητές για το σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα να επιμείνω σε τέσσερα σημαντικά μηνύματα που προέκυψαν και από τη συζήτηση και από την έκθεση. Το πρώτο θέμα είναι η σημασία που έχουν η καινοτομία και η έρευνα για τον τομέα των μεταφορών. Όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, γιατί οι μεταφορές είναι από τους σημαντικούς τομείς όπου έχουμε ηγετική θέση στον κόσμο χάρη στην καινοτομία μας, αλλά είναι και θέμα πολιτικής. Και δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές έχει σημαντικ... αφιερώνει σημαντικό τμήμα στο θέμα της καινοτομίας και της έρευνας, που θεωρούν αναπόσπαστα στοιχεία του τομέα των μεταφορών. Είχαμε τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τον ορίζοντα του 2020 και το πρόγραμμα για την έρευνα στις μεταφορές. Μην ξεχνούμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το κεφάλαιο των μεταφορών όταν κάποιοι συνάδελφοι ακόμη και εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσπαθούν να το περικόψουν. Δεύτερο σημαντικό θέμα που προκύπτει από την ανάγνωση της έκθεσης είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών και των ε, ερευνητικών πρωτοβουλειών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως και είμαστε υπερήφανοι γιατί ε, στις μεταφορές προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία, ε, την έρευνα μάλλον σημαντικό μέσο διαμόρφωση των πολιτικών. Αυτό ισχύει για την πολιτική του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, του ΣΕΖΑΡ και την προσπάθεια να δώσουμε στον τομέα μια πραγματική ισχύ με την έρευνα και την καινοτομία και επίσης έχουμε προωθήσει πολιτικές που προάγουν την καινοτομία. Και η τελευταία πρωτοβουλία που σας υποβάλαμε είναι η πρωτοβουλία για τις μεταφορές όπου λάβαμε υπόψη τα, τις νέες εξελίξεις, τις τεχνολογικές, τα νέα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα και υποβάλαμε και νομοθετική πρόταση ώστε τέτοιου είδους ε, μεταφοράς να ενταχθούν κανονικά στην αγορά. Τρίτο σημαντικό θέμα είναι η σύσταση του εισηγητή να εξετάσουμε μία σειρά θεμάτων και να έχουμε μία πιο σφαιρική προσέγγιση, δηλαδή να μην επικεντρωθούμε μόνο στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υφιστάμενων οχημάτων, αλλά να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτά τα οχήματα ή πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Και υπάρχει έκκληση στην έκθεση να είμαστε πιο δημιουργικοί και το θέμα του συστήματος μεταφορών να το ε, θεωρήσουμε να το εξετάσουμε υπό διαφορετική σκοπιά. Επίσης, ε, να γίνει καλύτερη εσωμάτωση των υποδομών στις μεταφορές, γιατί μερικές φορές αποσυνδέουμε τα οχήματα από τις υποδομές. Και το μήνυμα της έκθεσης είναι πολύ χειρό να συνδυάσουμε τις, μεταφορές με τα οχήματα τις υποδομές με τα οχήματα, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο θέματα, έχουν σχέση οι υποδομές με τα νέα ε, οχήματα. Και Θέλουμε ευφυή συστήματα μεταφορών. Και τέλος, περισσότερη ολοκλήρωση μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών τομέων. Είχαμε το πρόσφατο παράδειγμα με την πρωτοβουλία Smart Cities, ευφυής πόλης. Εκεί θέλουμε να αναπτύξουμε ενέργειες μεταξύ των μεταφορών, της έρευνας μεταφορές, της έρευνας της τεχνολογίας επικοινωνίας και της έρευνας στην ενέργεια. Και τέταρτο σημαντικό μήνυμα της έκθεσης είναι ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα όλο το πλωστάσιο των μέσων μας. Και έχουμε αρκετά μέσα στη διάθεσή μας. Έχουμε επίβολα σχέδια, σημαντικές συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες τα τελευταία χρόνια. Και επίσης και κοινωνικο-οικονομική έρευνα, πιο ήπια μορφή έρευνας, που είναι πολύ σημαντική για να αντιληφθούμε καλύτερα τις ανάγκες των νέων μέσων μεταφοράς και επίσης να συγκεντρώσουμε τα κατάλληλα στοιχεία για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις με τις πολιτικές μας. Εν λοιπόν, η έκθεση αυτή αφορά την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που παρουσιάζει μια στρατηγική άποψη για τις μεταφορές και μια πιο, ένα πιο μακροχρόνιο ε, ορίζοντα. Αργότερα θα υποβάλουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις στα πλαίσια του ορίζοντας 2020 και για την επόμενη επταετία των δημοσιονομικών προοπτικών και από αυτήν την άποψη η έκθεση θα συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση και αυτών των προτάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάικλ. Ναι, ευχαριστώ ε, για τα σχόλια όλα. Ε, θα απαντήσω σε ορισμένα μόνο, αλλά να πω ε, ότι έχουμε περιορισμό στην έκθεσή μας, ε, στον όγκο, ε, στους χαρακτήρες. Γι' αυτό δεν μπορούσα να τα βάλω όλα στην έκθεση. Γι' αυτό υπάρχουν και τροπολογίες και εμείς θα κάνουμε έξτρα τροπολογίες για να ε, μπορέσουμε να υπερβούμε αυτό το όριο. Για τον κύριο Πίρκερ να πω που τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι πόλεις. Μα εκεί είναι ακριβώς τα προβλήματα. Το 70% των εκπομπών όχι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα, γιατί αναφερθήκατε και στα οξίδια του αζότου, στα νόξ, ε, είναι στις πόλεις. Ακριβώς, αν δεν το λύσουν οι πόλεις αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί πουθενά. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να κινηθούμε. Και στο Φερολίνο, ε, ε, εδώ και 18 χρόνια δεν έχουν αλλάξει ε, οι ε, τιμές ε, στους χώρους στάθμευσης, στα πάρκινγκ, ενώ έχουν πολλαπλασιαστεί τα εισιτήρια του προαστιακού σιδηροδρόμου, ας πούμε. Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες προώθησης, είναι σημαντικό αυτό μεν, αλλά είναι ένα από τα πέντε μειονεκτήματα. Άλλο είναι ο θόρυβος. Μόνο σε χαμηλές ταχύτητες ε, επηρεάζεται αυτό. Είναι πολύ πιο σημαντικό εκεί το οδόστρωμα και τα ελαστικά. Επίσης, το κόστος. Κάθε αυτοκίνητο ε, χρηματοδοτείται κάθε χρόνο με 1.600 ευρώ έχει υπολογιστεί αναφορολογούμενο. Ε, λοιπόν, δεν είναι μόνο ο κινητήρας ε, να βελτιωθεί, αλλά και τα οδοστρώματα και τα ελαστικά. Ε, είναι γενικότερο το ζήτημα για την προστασία του κλίματος. Για τον κύριο Λιμπεράτσκι. Τον ευχαριστώ για την κοινωνική διάσταση που υπογράμμισε. Το κάναμε, το κάνατε κι εσείς κύριε ε, ίσως ε, πολύ συνοπτικά. Περιμένω με ενδιαφέρον και τις τροπολογίες σας. Η χορύπανση, ο θόρυβος ε, αναφέρθηκε επανειλημμένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που αγωνίζονται όλες οι πολιτικές ομάδες για το θόρυβο, πολύ συγκεκριμένα. Ε, θα βρούμε μια πολύ ωραία συμβαστική τροπολογία για να μας καλύπτει όλους. Κυρία Μπιλμπάο, συμφωνούμε πολλά ε, με, με ένα διαφωνή, λέει η κυρία Μπιλμπάο, για τον ανταγωνισμό και τις διάφορες δομές. Βεβαίως μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση, να δούμε τι τροπολογίες θα κάνετε και τι συμβιβασμούς θα ε, βρούμε. αυτά τα τρία ίντερ που λέτε, δια ε, κινητικότητα, δια λειτουργικότητα, δια τροπικότητα, όλα αυτά τα ίντερ να τα ξαναγράψουμε. Εγώ συμφωνώ και με την κυρία Ρόσπαχ. Για τον κύριο Κόχλιτσεφ, ε, για τα, για τα ποδήλατα έχουμε τώρα αυτά λεγόμενα e-bikes ε, και ανθεί αυτός ο κλάδος σε όλη την Ευρώπη χωρίς ούτε ένα σεντ κρατικά χρήματα θα μπορούσαν να αντιγράψουν τα αυτοκίνητα αυτά που γίνονται στα ποδήλατα. Δισεκατομμύρια δίνουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία για τα αυτοκίνητα, για το ποδήλατο. Ανθεί πραγματικά αυτός ο κλάδος. Και ε, η διαφορά τώρα για τα υψόμετρα και ποιος έχει λόφους και ποιος έχει ίσωμα και επίπεδες επιφάνειες. Αυτό το e-bike που έχει εφευρεθεί είναι πάρα πολύ ωραίο ποδήλατο και δεν χρειάζεται καθόλου κρατική ενίσχυση. Το θέμα ε, για τα τροχέα, η κυκλοφοριακή αγωγή δεν θα πρέπει να ε, έχει ως επίκεντρο μόνο τα θύματα από τροχέα, αλλά και τους θύτες, τους οδηγούς δηλαδή. Ε, Το Βερολίνο για τρίτη φορά διεξήχθη πρόσφατα μια έκθεση για ποδήλατα, Βέλο Μπερλίν. <laughs> Από παλιά αυτοκίνητα ανακυκλώθηκε ε, η Λαμαρίνα και ε, έχουν φτιαχτεί πλέον ποδήλατα. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ανακύκλωση που επιδείχθηκε σε αυτή την έκθεση εκεί και βλέπουμε πώς μπορεί να αυτοκίνητο να τελειώσει τον κύκλο του. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την συνεργασία και για τα όσα είπε. Βεβαίως η ε, ολοκληρώση και τα μεγαλεπίβολα ερευνητικά προγράμματα είναι ωραία και καλά, ε, αλλά και δεν διαφέρουμε πολύ στις απόψεις μας, μπορούμε να βγάλουμε μια καλή έκθεση και τέλος να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη γραμματεία μας και τους συνεργάτες μου και τους κοιόδης συγητές. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Kramer. Can I just remind... Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Να σας υπενθυμίσω την προθεσμία για την κατάθεση των απολογιών ε, για την έκθεση που περιμένει ανυπόμονα ο κύριος Κράμερ λίγη στις 9 Απριλίου. Η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή μας στις 18 Ιουνίου. 9 Απριλίου λοιπόν ε, είναι η διορία για τις τροπολογίες και 18 Ιουνίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, Ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Eurocontrol, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού δηλαδή για την ασφάλεια της ε, αεροναυτιλίας. Ο συγγετής μας είναι ο κ. Κόχλιτσεκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι το αεροκοντρόλ, οι δραστηριότητες του αεροκοντρόλ είναι, είναι κάτι που ε, χρησιμοποιούμε όλοι γιατί ταξιδεύουμε πολύ, είμαστε πολύ συχνοί επιβάτες ε, αεροπλάνων και βλέπουμε ότι μερικές φορές υπάρχει συμφόρηση και στις αεροπορικές μεταφορές. Έχουμε και το σχέδιο ΣΕΖΑΡ που θα είναι ε, ανεκτήμητης σημασίας στο σχέδιο για τους Ευρωπαίους, ε, ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες, για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και με τον συνάδελφο Γεζεμπόφσκι είπαμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη κατάσταση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εναέριων μεταφορών και επίσης να προσδιορίσουμε κατά πόσο η αρμόδια, ο αρμόδιος οργανισμός για την ασφάλεια στην αεροπλοεία έχει αρκετές μεταφορές. Η διαχείριση των αερομεταφορών είναι περίπλοκος κλάδος και εξελίσσεται ραγδαία. Και τα περισσότερα κράτη-μέλη, με εξαίρεση την Εστονία, όλα, όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση την Εστονία, συμμετέχουν και στη Eurocontrol. Οπότε μας ενδιαφέρει μία συμφωνία που θα προσδιορίζει με σαφήνεια το ρόλο της Eurocontrol, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Ενεργοαυτελείας θα είναι ο ενιαίος φορέας για την εφαρμογή και του Ευρωπαίου, ενιαίου Ευρωπαϊκού Ορανού και επίσης προσδιορισμός των ε, αρμοδιοτήτων της Eurocontrol σχέση με την ΕΑΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της, ε, των Αεροπορικών Μεταφορών. Έχουμε δύο ε, δυνατότητες ως προς την έκθεση, να δεχτούμε την συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Eurocontrol, ή να την απορρίψουμε. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε αυτή την ε, συμφωνία. Ευχαριστώ κύριος Δεγκράντες Πασκόλ εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Σιγητά, κύριε Κόλιτσεκ. Δεν είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή, γιατί αυτή τη στιγμή διαδικαστικά ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζεται στην αποδοχή ή στην απόρριψη τη συμφωνία. Και δίκιο έχει ο εισηγητή που μας συστήνει να εγκρίνουμε την έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Eurocontrol. Είναι αναφυσβήτητο αυτό. Γιατί. Καταρχήν ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ του Eurocontrol και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα προσδιορίζονται τα διάφορα επίπεδα συνεργασίας που από το δημιουργούν μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων φορέων ελέγχου τη ενέργεια κυκλοφορία και εξασφαλίζουν ασφάλεια στου ευρωπαϊκού εθέρε. Δημιουργείται μια μεικτή επιτροπή ε, από εκπροσώπους και των δύο μερών που θα συνέρχεται άπαξ το χρόνο για να αναλύουν και να εξετάζουν τους στόχους του, της Eurocontrol όπως περιλαμβάνονται και περιγράφονται στην έκθεση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης των αεροπορικών μεταφορών που θα είναι ολοκληρωμένο, θα ε, εξασφαλίζει ασφάλεια, αποδοτικότητα, προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά προς όφελος των επιβατών ε, και των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης προσπαθούμε με την έκθεση αυτή να δώσουμε την απαραίτητη όθηση για την εφαρμογή του, Ευρωπαίου, ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού εξασφαλίζει το συντονισμό των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε επίση με τον εισηγητή που προτείνει έγκριση της έκθεσης, έγκριση συγγνώμη τη συμφωνία αυτή. Οπότε θα πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και οποιαδήποτε τέτοια πρόταση είναι ευπρόσδεκτη. Με βάση το άρθρο 81 του κανονισμού η δική μας αρμοδιότητα είναι να δεχτεί ή να απορρίψει την συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να εγκρίνουμε την συμφωνία αυτή, τηρώντα και τη σύσταση του εισηγητού μα με τον οποίο συμφωνούμε απόλυτα. Ο κύριος Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, όταν συζητούμε για την αεροναυσιπλοεία, για αεροναυτιλία, θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ευρώπη ανήκει σε εκείνου του τομεί που είναι πιο κινητοκοποιημένοι και ενοποιημένοι και ολοκληρωμένοι. Έχουμε ένα κοινό πλαίσιο, ένα κοινούς εθέρες, αλλά Ακόμα δεν έχουμε ε, κοινέ ε, δυνατότητες ρύθμισης και κοινού κανόνες. Και εν μέρη αυτό μας περιορίζει και δεν έχουμε επιτυχία ε, στη δράση μας. Τώρα, τίθεται το εξής ερώτημα. Θα πρέπει αυτή τη συμφωνία να τη δεχτούμε και θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να το εξετάσουμε. Βέβαια στις λεπτομέρειες μπορεί να είχαμε άλλα κέντρα βάρους, άλλες προτεραιότητες, αλλά πιστεύω ότι αυτό για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες χρειάζονται πιο μαζικά βήματα να γίνουν, αλλά δεν είναι τώρα η δουλειά μας αυτή. Αυτό που καλούμαστε να πούμε είναι ένα ναι ή ένα όχι, αν θα δεχθούμε ή αν θα απορρίψουμε τη συμφωνία. Εδώ συμφωνώ λοιπόν και με τον εισηγητή και με τον πρόλα Λίσαντα, τον κύριο Γκράντες Πασκουάλ και συμφωνώ να εγκρίνουμε τη συμφωνία και την έκθεση του κυρίου Κόχλητσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπεργκε. Ευχαριστώ πολύ. Σε γενικές γραμμές μπορώ και εγώ να συμφωνήσω με τη βαρούσα έκθεση στους ενιαίους ε, ευρωπαϊκούς εθέρες δεν προχωρεί η υπόθεση, αλλά αυτό δεν είναι επειδή φταίει η Eurocontrol, αλλά τα κράτη-μέλη είναι εκείνα ε, τα οποία με μεγάλη χαρά εξαγγέλουν αυτούς τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Αλλά όταν ε, τους φεύγει η αρμοδιότητα από τα χέρια, ε, σε κάποιο τμήμα λειτουργικό του ουρανού, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Ε, σε πολλούς ε, τομείς παρατηρείται αυτό, ότι μας αρέσουν οι ωραίες εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια, αλλά όταν θίγονται εθνικά συμφέροντα, Βέβαια αυτό ελέγχεται πιο το ορίζει, γιατί καμιά φορά εθνικό συμφέρον είναι και οικονομίες. Ε, ε, τότε ε, ε, όλα είναι πάρα πολύ επίπονα, χρονοβόρα και δυσάρεστα. Τώρα, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να δούμε πού υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ ΆΣΑ και Eurocontrol. Γιατί εμένα θα με δυσαρεστούσε πάρα πολύ να πληρώσει την ύφη μόνο του Eurocontrol. Γιατί σε πολλούς τομείς, στην ΕΑΣΑ που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών, ε, υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί και ζητούν πράγματα τα οποία ζητάει και ο κλάδος των αερομεταφορών. Δηλαδή κάπως ευθυγραμμίζεται. Και εκεί χρειάζεται άλλη τακτική να έχει ε, λόγο και αποφασιστικό Eurocontrol και να μην λύνονται ε, προβλήματα σύγκρουση αρμοδιοτήτων όλα προ όφελο της ΕΑΣΑ. Γιατί υπάρχει ένας παραλληλισμός, μια ταύτιση συμφερόντων που θα πρέπει να διασκεδαστεί. Κύριε Φώστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εισηγητές. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια Νομίζω ότι είναι αρκετά επεξηγηματική η ίδια η διατύπωση και μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ είμαι υπέρ του αεροκοντρόλ. Νομίζω ότι έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια στα πλαίσια της διαχείρισης των μετακινήσεων και το ότι υποστήριξαν τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς και την επιτυχία που τους χαρακτήρισε είναι ένα τεχνολογικό θα έλεγα <clears throat> ακατόρθωμα. Βέβαια θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πώς έχουν τα πράγματα. Αντέδρασαν αρκετά γρήγορα όταν είχαμε το πρόβλημα με την ηφαιστειογενή, με το σύννεφο από τα ηφαίστεια της Ισλανδίας και θα πρέπει επίσης να τιμήσουμε εδώ και τον τελευταίο Γενικό Διευθυντή, τον David Μακμίλαν που δεν είναι πια εκεί, και ο οποίος προώθησε γενικά την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης. Θα ήθελα να με διαβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξής. Προφανώς θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο νέος γενικός γραμματέας τους, ο Πατεχή, ο οποίος ήταν υπεύθυνο για το ΣΕΖΑΡ, <clears throat> θα αναλάβει το Σεπτέμβριο και ελπίζω ότι αυτό να μην, δεν θέλω να θίξω τις παρούσες υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται. Ασχολείται με το Σεζάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Και εδώ ο ρόλος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντικός έτσι ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις, να μην υπάρχουν επαναλήψεις, να μην υπάρχουν περιττοί ανταγωνισμοί οι οποίοι χαρακτηρίζουν μερικές φορές ε, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Μάθιου ξέρει γιατί μιλάω. Θέλουμε τα πράγματα να πάνε καλά. Μία μικρή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να μου δώσει κάποιες περιορισμένες πληροφορίες για τα μέλη της ειδική Επιτροπής στα άρθρο 4. Και ποιοι είναι τα μέλη της Μικτής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Baldwin από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much. I can be very brief, uh, Θα είμαι σύντομο Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη σωστή συζήτηση υποστηρίζοντας αυτή τη σημαντική συμφωνία για την κυρία Λίχτενμπεργκερ και την κυρία Φώστερ και για τα σχόλιά τους. Να πω ότι είμαστε επίσημα μέλη και εμείς της ομάδας υποστηρικτών του Eurocontrol. Πράγματι και υπό την καθοδήγηση του Μακμίλαν και με τους νέους υπεύθυνους τα πράγματα πάνε πολύ καλά μεταξύ μας. Κυρία Φώστερ, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι ακριβώς να διασφαλίσουμε την απουσία της επικάλυψης και να δημιουργήσουμε συνέργειες με το Eurocontrol. Και το Eurocontrol ε, επιβεβαιώθηκε η θέση του για μια ακόμη φορά σαν το τεχνοκρατικό κομμάτι και επιστημονικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια την οποία κάνουμε στον τομέα των αερομεταφορών σχετικά με τις κοινέ επιτροπές. Περιλαμβάνει εκπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ιδίου του Eurocontrol και καλούμε φυσικά εμπειρογνώμονες όποτε αυτό χρειάζεται. Η μεικτή Επιτροπή θα συνεδριάσει το τέλος του μηνός Απριλίου και ήδη ελπίζουμε σε αυτή την πρώτη συνάντηση να υπογράψουμε τρία παραρτήματα ή τρία προσαρτήματα και για την ασφάλεια των αερομεταφορές, στις αερομεταφορές και σε σχέση με τη συνεργασία με τις στρατιωτικές αρχές. Πρόκειται για μια ζωντανή συμφωνία, ζώσα συμφωνία, ενδιαφέρουσα η οποία δεν προορίζεται για τα αρχεία. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί σας όποτε το επιθυμείτε. ανήκει έτσι κι αλλιώ στην Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Eurocontrol. Κύριε Κόχλιτσακ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι ήδη εκφράστηκαν θετικά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και εγώ για την συνεργασία με όσους βοήθησαν στην προετοιμασία. Θέλω να ευχαριστήσω τους βοηθούς μου, δεν χρειάζεται κάποιο άλλο σχόλιο. Προσωπικά θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την Εσθονία, λέει ο κ. Κόχριτσεκ, και γιατί δεν συμμετέχει στο Eurocontrol. Αλλά είναι περιθωριακό το συγκεκριμένο θέμα, γιατί το μέγεθος της χώρας και η, ζώνη που καλύπτει είναι ε, σχετικά μικρή. Ίσως να εξοικονομούν χρήματα, όπως ακριβώς έκανε και με τον δικό της ενέργειο χώρο η Τσεχία. Πράγματι αυτό δεν σταμάτησε. Δεν σταμάτησε τις χώρες να παίρνουν μέρος στο Eurocontrol στο παρελθόν και το ίδιο θα γίνει ελπίζω και με στην Εστονία. 4η Απριλίου Τετάρτη μόνη τροπολογία που μπορείτε να προτείνετε είναι να απορριφθεί η συμφωνία αλλά εγώ είμαι θετικός εκφύσεως και γι' αυτό δεν ήθελα να πω ότι η προθεσμία σας για την απόρριψη είναι η 4η Απριλίου, αλλά περί αυτού πρόκειται στην πραγματικότητα. Και φτάνουμε στο τέλος σε αυτή τη φάση αυτού του τμήματος. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 23 Απριλίου. Φτάνουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, στο τέλος, και ο Σίμψον, για τη συνεδρίασή μας. Θα επανέλθουμε αύριο ή στα 9 για να ψηφίσουμε. Παρακαλώ να πάρετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες μαζί. Τέλος.